Παρακαλώ οι συνάδελφοι που έχουν κάτι άλλο να κάνουν, ας το κάνουν εκτός εθούσης, για να συνεχίσουμε και εμείς να περάσουμε στο επόμενο σημείο για τις παγκόσμιες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον κύριο Ενέκο Λανταμπούρο από το Ίδρυμα Νότχο Εγώπ και τον κύριο Κέβιν Βάτκινς ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Think Tanks. με αφορμή τη δημοσίευση μελετών με θέματα συμμετοχή της Ευρώπης στον κόσμο και προσοχή σε αυτό που θα πω είναι τεράστιος ο τίτλος γιατί τα προβλήματα της Ευρώπης χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις και τα προβλήματα του κόσμου απαιτούν ευρωπαϊκή δράση αντιστοίχως. Θα ακούσουμε τους κυρίους Λανταμπούρου και Βάτκινς 10 λεπτά έκαστος και κατόπιν ερωταπαντήσεις. Καλωσορίζω τον κύριο ε, Γκρέβι Σόλσε Λαπόρτ από το Ευρωπαϊκό Think Tank. Αν είναι εδώ, καλωσορίσατε. Κύριε Λάντα Μπούρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το δύσκολο και λεπτό καθήκον που αναλαμβάνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παγκόσμια πραγματικότητα απαιτεί ένα ε, ρόλο ε, ακόμη πιο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το παρελθόν. Το διακύβευμα είναι η παρουσία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Το ε, Ινστιτούτο Jacques Delors είναι ένα think tank. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων μας ο πολίτης και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια Ο ανταγωνισμός και η αλληλεγγύη και η συνεργασία, θέματα προσφυλής στο Ζακ Τελόρ, στο ρόλο του ως κινητήρης δυνάμεις ε, της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης και τρίτος άξονος, εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι στο Think Tank μας έχουμε αποδώσει τη δέουσα σημασία στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μας διακρίνει από άλλα θεσμικά όργανα και αντίστοιχα think tank είναι πως ενώπιον των προβλημάτων επιθυμούμε να μην είναι θεωρητική ή δογματική η προσέγγισή μας, αλλά ε, κατά κύριο λόγο ρεαλιστική. Ε, ο στόχος ε, ενό think tank είναι να υπηρετεί τους ε, ηθήνοντες, αυτούς που μετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, τους βουλευτές, να συμβάλλουμε στον προβληματισμό. Σακ όπως παραδείγματο χάρη στο Ζακ Τελόρ, στον κύριο Γκικού, ε, σε μια σειρά από ανθρώπους που έχουν ε, στο παρελθόν λάβει πολύ σημαντικέ αποφάσεις ε, για το μέλλον της Ευρώπης και σε σχέση με άλλα think tank που επίση επιτελούν ένα σημαντικότατο έργο στην Ευρώπη, αυτό που μας διακρίνει ότι αποφασίσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μα σε μια σειρά από προτεραιότητε που εμεί κρίνουμε ω απαραίτητες ε, και σε σχέση με τις οποίες κρίνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόοδου ε, στο μέλλον, κατά αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Εξού και η σημασία ανταλλαγής απόψεων με εσάς, που καλείστε να υπομειστείτε την ευθύνη που σας αναλογεί και να συμβάλλετε στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη βάση παρελθούς εμπειρίας μας αποφασίσαμε να εκπονήσουμε πριν διεξαχθούν οι ευρωπαϊκές εκλογές ένα μανιφέστο. Ανάληψη δέσμευσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, τυκλοφορείτο και εκεί ε, ε, παραθέσαμε τις προτάσεις μας. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, στην αρχή μας υποσχεθήκατε 15 λεπτά, τώρα μου είπατε 10, ελπίζω να μην με ξαναδιακόψετε και να μου δώσετε μόνο 5 λεπτά, θα περάσω στην ουσία. Μην με προκαλείτε, λέει ο Πρόεδρε μου. Λοιπόν, ε, επί της ουσίας. Είναι μάλλον ε, τετριμένη αυτή η παρατήρηση, αλλά ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρώπη, τα κράτη-μελή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απολέσει σε έναν ορισμένο βαθμό την επιρροή τους στη διεθνή σκηνή τόσο ε, σε πολιτικό, οικονομικό αλλά και δημογραφικό επίπεδο. Αυτό ε, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να βασίσουμε τις σκέψεις μας ε, σε αυτό. Δεύτερον, έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στον κόσμο, κυρίως ε, στη, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Νότο ε, και προς την Ανατολή. Είναι καυτή η επικαιρότητα και λίγα ανησυχητική. Υπάρχουν ε, δύο στοιχεία που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε υπάρχει, χρειάζεται, μια, χρειάζεται να αντιδράσουμε, χρειάζεται να αναλάβουμε νέα δέσμευση στην ε, Ευρώπη για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, παρακμή που φαίνεται αναπόφευκτη και αφετέρου για να σταθούμε στο ύψος της νέας πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. διαπιστώνουμε σε αυτό το μανιφέστο που σας στείλαμε ότι κανένα ε, κράτος μέλος, ε, ανεξαρτήτως σημασίας, δεν είναι σε θέση από μόνο του να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις και να ε, προσφέρει λύσεις ε, στα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής που τίθεται για το ίδιο. Είτε πρόκειται για ειδικά ζητήματα όπως η Αραβική Άνοιξη, παραδείγματο χάρη η πολιτική του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία, είτε πρόκειται για γενικότερα πιο οριζόντια ζητήματα, δεν ναι. ε, υπάρχει δυνατότητα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή να έχουν την δέουσα επιρροή ώστε να επηρεάσουν αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους. Ένα κόσμο λοιπόν που ή γίνεται όλο ένα και ανταγωνιστικότερος και, ε, όπου πολλαπλασιάζονται αναμφίβολα οι διενέξεις. γινεται ολοένα και ανταγωνιστικοτερος διάσταση είναι ε, εκ των ουκ άνευ για να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε δράση. Το θέμα είναι να προσδιορίσουμε την ε, προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πλαίσιο που παρουσιάζει τόσο μεγάλες δυσκολίες. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί. Πριν από λίγα χρόνια είπε ο Ζακ Ντελόρ με ξεκάθαρο τρόπο πώ χρειάζεται διανοητική και πολιτική ορίμανση για μία σειρά ετών, ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε μία τέτοια εξωτερική πολιτική. Πόρο απέχουμε από κάτι τέτοιο και χρειάζεται σε ε, θεωρητικό, διανοητικό και σε πολιτικό επίπεδο πολλής χρόνος ούτως ώστε να ρίξουμε τα θεμέλια μιας τέτοιας εξωτερικής πολιτικής. Ε, δεν μπορούμε δεν να παραβλέψουμε ε, το γεγονός ότι προσπαθώντας να επιταχύνει τη διαδικασία απέτυχε το Μάστριχ, Η συνθήκη του Μάστριχ είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και έθετε μία σειρά στόχων για να εξασφαλίσει ακόμη και σε αμυντικό επίπεδο τη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδύνευσε σε μεγάλο βαθμό και παρότι σημειώθηκε μεγάλη πρόεδρος και παρότι το Δεκέμβρη το τελευταίο Συμβούλιο των ε, Υπουργών Αμήνης καθώς και το ε, Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ε, διερεύνησαν το μίσο όπου θα μπορούσαμε να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο. Σφαιρικά θα έλεγα ότι αυτοί που συνέταξαν τη συνθήκη είχαν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Απέχουμε πάρα πολύ από το στόχο που είχαν θέσει. Υπάρχει ε, υπάρχουν αντιφάσεις, μεγάλες αντιφάσεις και διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Όλοι έχουν διαφορετικό παρελθόν, κυρίως μεγάλες χώρες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία έχουν τέτοιο παρελθόν, τέτοια ιστορία, ώστε δυσκολεύονται να καταλήξουν σε ένα κοινό παρονομαστή για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ε, το εξίσου σημαντικό ε, και ανησυχητικό σε αυτή τη διαπίστωση που κάνω κατά τη γνώμη μου είναι η έλλειψη φιλοδοξίας των ε, ηθινόντων, κάτι που χρειάζεται για να προοδεύσουμε περισσότερο, είτε διότι δεν μπορούν, είτε διότι δεν θέλουν οι ηγέτες των ε, μεγάλων χωρών δεν έχουν αυτή τη βούληση. Ίσως ε, με τα πρόσφατα γεγονότα θα αντιληφθούν ότι θα πρέπει να ενωθούν για να αντιδράσουν καλύτερα ε, και να αντιδράσουν σε σχέση με τις εισαγωγικά απειλέ. Ίσως, ίσως γίνει και αυτό. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να πούμε όχι, δεν γίνεται, ε, ε, να αφήσουμε την ητοπάθεια να μας νικήσει. Όχι, και γι' αυτό στείλαμε αυτό το μανιφέστο ε, για την τρέχουσα θητεία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε την δράση σε πέντε διαφορετικούς τομείς για να ε, δρομολογήσουμε μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ε, μόνο ευκταίες αλλά τις οποίες κρίνουμε ότι είναι πολιτικός πώς εφαρμόσιμες. Αυτό είναι το σημαντικό. Το δεν έχω χρόνο και θα ε, είμαι ε, πάρα πολύ γρήγορος. Εξάλλου σας παραβεύω στο έγγραφο που σας έχουμε ήδη στείλει. Λοιπόν, Ποιοι είναι το μίσο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σημειωθεί η πρόοδος. Προετοιμασία της διαχείρισης των κρίσεων, ενίσχυση των ε, αμυντικών ικανοτήτων, των ικανοτήτων μας και ικανοτήτων λήψη λήψης συλλογικών αποφάσεων. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μιλήσαμε για τη συνεργασία για τα μη επανδρομένα Μιλήσαμε για τη δρομολόγηση της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων. Υπάρχουν, υπάρχουν στοιχεία σύγκλησης σε αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν που αξίζουν να εξεταστούν περαιτέρω ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Στον τομέα της κοινή αμήνης ε, είναι επιτακτική ανάγκη κατά τη γνώμη μας ε, να είναι ε, ισχυρή ε, και συνειδητοποιημένη η θέση μας σε σχέση με κάποιες γεωγραφικές οντότητες και χώρες, όπως η Ρωσία, Είναι θέμα επιβίωσης, ε, θα πρέπει να είναι κρατεότερη η θέση μας για να μπορέσουμε, εάν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας. Πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική ασφάλεια Όμω κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Είναι σημαντικό ε, το έγγραφο που ε, είχε καταρτιστεί όταν ήταν στον Άτομο Χαβιέ Σολάνα Νομίζω ότι η νέα ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει να σπεύσει ώστε να αναθεωρηθεί και να επαναπροσδιοριστεί η πολιτική ασφάλειας αναλύοντας ε, την τωρινή πραγματικότητα και τις απειλές ε, που έχουν στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να μπορέσουμε σχέση με αυτές τις απειλές να προτάξουμε και εμείς μια απάντηση, να έχουμε μια συγκεκριμένη αντίδραση και θα έλεγα μάλιστα πώς ο θρησκευτικός ε, ριζοσπαστικισμός ε, και οι εκδηλώσεις του επιτόπου έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι ενδιαφέρει η κατάσταση σε σχέση με αυτή που αντιμετωπίζαμε πριν από μία δεκαετία. Και γι' αυτό ε, χρειαζόμαστε ένα προσδιορισμό της πολιτικής ασφάλειας μετά από προσεκτική ανάλυση της κατάστασης και έτσι μόνο θα ορίσουμε νέες προτεραιότητες και θα ξεκινήσει ε, ο απαιτούμενος πολιτικός διάλογος όχι μόνο σε σχέση με αυτές τις ε, χώρες και ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα θα διαδραματίσει ε, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τέλος για να μην μακρηγορώ σε αυτό το τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των κρίσεων δεν υφίσταται συγκεκριμένο μένο ε, εμπόδιο ώστε να αποφύγουμε ε, τη σύνταξη μιας λευκής βίβλου για την ε, ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βλέπουμε τα εξοπλιστικ... τους εξοπλιστικούς προϋπολογισμούς ανά τον κόσμο, βλέπουμε ότι είναι στάσιμοι ή μειώνονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαστολή με όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Ε, άρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική μα. Δεν λέω ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά είναι απαραίτητα. Θα ήταν ανεύθυνο από πλευρά μας ε, να μην αποπειραθούμε καν να ε, ξεκινήσουμε αυτή την άσκηση σύσταση λευκής βίβλου. σε ποιον άλλο τομέα μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στην ενεργειακή πολιτική, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ασφαλέστερη τροφοδοσία ε, και ο Ζακ Τελόρ ε, πριν από λίγα χρόνια είπε ότι η ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας όπως και η ΕΚΑΧ τη δεκαετία του 50 θα μπορούσε να αποτελέσει απαραίτητο στοιχείο για να τονώσουμε τον ανταγωνισμό, να ανταποκριθούμε στις μεταβολές του ενεργειακού τοπίου και να ανταποκριθούμε στις νέες και αυξημένες απαιτήσεις των αναγκών μας ως προς το φυσικό αέριο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της Ρωσίας σε, αυτό το, αυτή τη σκηνή. Ε, βλέπουμε ότι χρειάζεται βεβαίως η εσωτερική ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέραν αυτού σε διεθνές επίπεδο ο, η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να συνάδει, να συμμορφώνεται με τους στόχους μας. Θα πρέπει επίσης ε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ε, κυρίως ο Πρωθυπουργό Ντόναλτ Τάσκα που σύντομα θα αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο οποίος είχε υποστηρίξει αυτή την πρόταση του Ζακ Ντελόρ, είχε ο ίδιος πει πως σε αυτή τη θητεία ακριβώς θα μπορούσε αυτό να είναι σημαντική πρόοδος, να έχει σημαντικές επιπτώσεις και κυρίω να γίνει αντιληπτική αυτή η πρωτοβουλία από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό ήταν ο δεύτερο τομέας. τρίτο τομέας τώρα. Πρόκειται για τους ε, σημερινούς και μελλοντικούς ανθρώπινους πόρους ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, μεταναστευτική πολιτική μας. Ως εκ τούτου είναι ε, απαραίτητο να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Βιώνουμε δράματα καθημερινά λόγω των νέων δεδομένων σήμερα η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει ασφαλέστερα τα σύνορα και να αναχαιτήσει τη λαθρέα μετανάστευση. Δεν μπορούμε να έχουμε μια μεταναστευτική πολιτική που εστιάζεται ε, ε, υπερβολικά σε αυτή αυτές τις ε, ε, πτυχές ε, της ασφάλειας. Σημαντικό είναι αυτό, αλλά υπάρχει μια σφαιρικότερη πρόκληση, μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να υπομισθούν το βάρος της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής καταπολέμηση αυτής της οδυνηρής πραγματικότητας ε, της παράνομης μετανάστευσης χρειάζεται κοινοτικοποίηση και αλληλέγγυα προσέγγιση των κρατών μελών με τρόπο ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον υφιστάμενο κίνδυνο αφενός αφετέρου πρέπει να ε, προβλέψουν την ε, γύρανση του πληθυσμού, τις νέες δημογραφικές εξελέξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαστούμε εργατικό δυναμικό σε λίγα χρόνια ε, και θα πρέπει να, με κάποια απόσταση και άρα και αντικειμενικότητα να αναλύσουμε την κατάσταση ούτως ώστε να υποστηρίξουμε, ε, να προωθήσουμε περισσότερο τη νόμιμη, ε, τη σύνομη μετανάστευση. Ναι, ναι και δεν θα μακρηγορήσω. Τέταρτος τομέας συνεργασίας, μάλλον δυνατότητας πρόοδου είναι η μπορική ο εμπορικός τομέας. Ε, εκεί μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρώπης, μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο τα σύνορά μας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε σχέση με τις αναδυόμενες χώρες. Οι εξαγωγικές δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ισχυροί σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό μας βάρος στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις και μην ξεχνάμε φυσικά την TTIP ε, είναι ε, κρίσιμη σημασία στη Διατλαντική Συμφωνία ε, η προσέγγιση των προτύπων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και τον ΗΠΑ αφετέρου θα μπορέσει να δώσει νέα δυναμική ε, στις συναλλαγές ε, και να τονώσει και την αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη. Έχει υποθεί πολλά και σε όλες τις σχετικές συζητήσεις αλλά πρέπει να το τονίζουμε και επίσης ε, είναι... το ίδιο πρέπει να κάνουμε και σε σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό βέβαια απαιτεί μεγαλύτερη φιλοδοξία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να παραμελούμε τον αυξανόμενο ρόλο της Αφρικής τον 21ο αιώνα. Τελευταίος τομέας που προκρίνουμε στην μελέτη μας είναι η αναθεώρηση ε, της πολιτικής μας σε σχέση με τις γειτονικέ χώρες. Και διαπιστώνουμε εδώ μία αποτυχία. Για δύο βασικούς λόγους. Αυτό αφορά και τις προσπάθειες προς Ανατολάς αλλά και προς Νότον γιατί το 2004 έγινε μια προσέγγιση και εγώ τότε που την ηγεσία του Ρωμανού Πόντι είχα αναλάβει αυτό το θέμα, τότε που ήταν πρόεδρο εκείνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε υιοθετήσαμε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να εξεύρουμε κάποιε λύσει για τι ε, χώρε που δεν θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση που βρήκαμε ήταν το να διατυπώσουμε κάποιο είδου ε, ε, προσφορά για να τις ε, ελκύσουμε. Δηλαδή έτσι θα, θα, αυτές θα εξισούντο, θα ε, ανεδέχονται το κεκτημένο παντού. Οπότε κάτι, κάτι πετύχαμε αλλά θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι προς Ανατολάς δεν ενδιαφέρονται όλε οι χώρες, προς νότον δε, με την ε, αραβική άνοιξη και όσα ακολούθησαν, έχει σταματήσει ελκυστική η Ευρώπη. Είναι, είναι, αυτό το πρωτομοσία. Δεν είναι πλέον ε, ελκυστική η Ευρώπη γιατί δεν αρκεί αυτή μα η προσφορά. Α, ναι, επαρκεί να πούμε ότι πρόκειται να σα βοηθήσουμε σε αναπτυξιακό επίπεδο και πρέπει να ανοίξουμε στα προϊόντα σα, στα σύνορά μα και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη κινητικότητα για να έρχεται εδώ κόσμο από εσά. Ε, αυτά όλα δεν αρκούν για αυτές τις χώρες για ιδεολογικούς, ιστορικούς, πολιτικούς λόγους δεν τους αρκούν αυτά. Επομένως αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε και το σούτο μάλλον καθώς βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια τεράστια επιδείνωση της κατάστασης σε κάποιες ε, χώρες, στη Μεσογείο όπως η Λιβύα ή όπως και η Συρία. είδατε τι έγινε προς Ανατολάς, ο ίδιο πρόεδρος ε, Πούτιν δεν δέχτηκε την εξομάλυνση των σχέσεων με τις χώρες εκείνες. Δεν έχουμε τώρα το χρόνο, εξήγησα το χρόνο που μου διατέθη, αλλά πρόκειται για μια επιτακτική αναγκαιότητα το να δούμε πώς θα αναθεωρήσουμε εκ βάθρων αυτή μας την πολιτική σε σχέση με τους γείτονες. Και πρότασή μου είναι το να έχουμε μια διαφοροποιημένη, τολμηρότερη, πιο γενναιόδορη προσέγγιση με τις χώρες εκείνες που δέχονται να προσεγγίσουν το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό μας πρότυπο. Οπότε να κάνουμε περισσότερα, ας πούμε το Μαρόκο ή την Ισία. Και εκείνοι που δεν θέλουν ε, να έχουν προνομιούχες σχέση με την ΕΕ, να τους θεωρήσουμε απλά τρίτες χώρες και να επικεντρώσουμε δηλαδή τις προσπαθίες μας και τα, τα, μέσα πολιτικής και έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι κατακλείδη λοιπόν Έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάληψης δράσης για να έχουμε πρόοδο και οπότε γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε προσπάθειες μέσα από όρους. Έτσι. και επομένω ο αρμόδιο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή θα πρέπει να, έτσι να σημειώσει πρόοδο. Αυτό προβλέπεται από τη συνθήκη, δεν προβλεπόταν πριν. Οπότε, κάθε μήνα, μια πενταετία, το ίδιο πρόσωπο πρόκειται να προεδρεύει τα συμβούλια των Υπουργών. Αυτός πρόκειται να κάνει τη στρατηγική εφαρμογή, συντονισμό. Τεράστιο έργο έχει να επιτελέσει. Και επίσης είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών προς τα έξω. Αυτός, ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορμόδιος, Γιατί οι κοινωνικές πολιτικές είναι ισχυρές για ανάπτυξη, ενέργεια, μεταφορές κλπ. Αυτές οι πολιτικές κάθε μία προχωράει με τους επιτρόπους. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με, με τον συντονισμό και ο αντιπρόεδρο, ο αρμόδιος, θα πρέπει αυτό να κάνει τον συντονισμό και άρα θα πρέπει να αναβαθμίσει φυσικά και την υπηρεσία εξωτερική δράση. και να πετύχουμε όλα αυτά και επίση τώρα το, το, το, ιστερόγραφο κατά κάποιο τρόπο θα σα σας πω ότι έχουμε τώρα τέτοιε τεράστιε προκλήσει έχουμε τόσα προβλήματα γύρω μας. Οπότε κύριοι και κυρίες βουλευτές, εδώ στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπείτε τον Ευρωπαϊκό λαό, τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους λαούς της Ευρώπης, οπότε έχετε αυτό το καθήκον του, ώστε να απευθυνθείτε στις χώρες, μέλη και να πείτε τι θέλετε, τι κάνετε, πώς πασχίζετε για μια πιο ισχυρή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική, που είναι κάτι το οποίο θέλει ο περισσότερος κομμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, καλή τύχη, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζω ότι θα τηρηθούν τα χρονικά όρια όπως σας παρεκάλεσα. Κύριε Βότνης. Θα κάνω ό,τι μπορώ και πρώτα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς. Είδα ότι είναι η πρώτη μέρα του σχολείου πάλι και είναι και η πιο δύσκολη. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, παρηγορηθείτε με αυτή τη σκέψη. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο και την Επιτροπή Εξωτερικών που ε, έρχεται σε επαφή με την ομάδα εργαστηριών ιδεών, Think Tank μια τέτοια συζήτηση αν την κάναμε προ 10 ετών θα μιλούσαμε κυρίως για βοήθεια και ίσως και λίγο για εμπόριο και επενδύσεις. Στην έκθεσή μας τώρα εμείς λέμε κάτι βέβαια για βοήθεια αλλά λίγα πράγματα και κυρίως η ατζέντα που μας απασχολεί στην έκθεσή μας έχει κυρίως σχέση με το φάσμα θεμάτων που καλύπτεται εσείς εδώ στην Επιτροπή σας σε διάφορους τομείς. Αυτό που νομίζουμε ότι απηχεί η έκθεσή μας είναι κάτι που ίσως σας φανεί προφανές, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το επαναλάβω. Δηλαδή ότι ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και δραματικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, με την μετατόπιση αυτών των τευτονικών πλακών του πλανήτη, εντό εισαγωγικών βέβαια, με την απόσταση μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών και με τις αποστάσεις αυτές δεν μειώνονται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει και συνέχεια των παλαιών προβλημάτων. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο που ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που πεθαίνουν από ασυτεία ή από ασθένειες σχετικές με την ασυτεία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα, βεβαίως η φτώχεια είναι ένα θέμα και της εξωτερικής πολιτικής αυτόνομο. Είναι όλο και περισσότερο σαφές για μας, εργαστήρια ιδεών δηλαδή της ανάπτυξης, ότι αυτά που αποκαλούσαμε προβλήματα ανάπτυξης παραδοσιακά, στην ουσία είναι προβλήματα ανασφάλειας, είναι προβλήματα διακυβέρνησης, χρηστής διοίκησης, είναι προβλήματα οικολογικά είναι προβλήματα που συχνά είναι κοινά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών. Να σας δώσω λίγα παραδείγματα. Το πρώτο τμήμα του υποτίτλου μας αναφέρεται στην ανάγκη που έχει η Ευρώπη από παγκόσμιες λύσεις. Ένα είναι ο ιός έμπολα άμεση απειλή για την δημόσια υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και δεν έχει άλλη λύση παρά μονάχα την συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων υγείας στην Δυτική Αφρική. Επομένως διεθνή συνεργασία. Επομένως προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτιών και απειλές που υφίστανται πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Άλλο, η κρίση της μετανάστευσης μέσα από τα νερά της Μεσογείου προς την Νότια Ευρώπη. Μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό ως θέμα μεθοριακό. Βεβαίως είναι εν μέρη πρόβλημα μεθοριακό. Ταυτόχρονα είναι και ζήτημα φτώχειας. Είναι το αποτέλεσμα σε ορισμένε χώρες προέλευση μεταναστών της κατάρρευσης του περιβάλλοντος, της οικονομίας, ανασφάλειας επίσης και επομένως και φτώχειας. Πάλι σε ορισμένες από τις χώρες αυτές μάλλον σε ορισμένα από τα θέματα αυτά δεν μπορεί να εξετάσει κανείς μια ευρωπαϊκή λύση εκτός πλαισίου διεθνούς συνεργασίας. Και αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της εκθεσής μας. Ο κ. Μπρόκ που βλέπω ότι μόλις επανήλθε μεταξύ μας ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχόλιο που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από συνάντησες με την Επίτροπο Γεωργίευα και μιλούσατε για την Ουκρανία θα σας παραφράσω λίγο αυτό που είπατε. Είπατε ότι πρέπει να ρίξουμε όλους τους πόρους και την ενέργεια των χωρών της Ένωσης στην υπεράσπιση των αξιών μας και τονίσατε την ανάγκη στρατηγικού συντονισμού στην προσπάθεια αυτή. Μα ακριβώς αυτό είναι και το πλαίσιο που εφαρμόζουμε εμείς στο ευρύ φάσμα θεμάτων που μας απασχολεί στην έκθεσή μας. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω το χρονικό πλαίσιο που μου δώσατε. Θα πω λοιπόν ποια είναι η πρότασή μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολιτικές, έχει τους οικονομικούς πόρους, έχει τα εργαλεία και τις αξίες που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστούν οι κοινέ παγκόσμιες απειλές, αλλά και για να εκμεταλλευτεί τις παγκόσμιες ευκαιρίες. Το δικό μας επιχείρημα είναι ότι η ικανότητα της Ευρώπης να προστατευτεί και να παρουσιαστεί στη διεθνή σκηνή τίθεται σε κίνδυνο από τις αποτυχίες των κυβερνήσεων. Έχουμε τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αποτυχίες των κυβερνήσεων που θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι το θεωρητικό και αφηρημένο, είναι πραγματικές αποτυχίες, παραλήψεις των κυβερνήσεων σε πραγματικούς τομείς πολιτικής. Εμείς δεν έχουμε εντοπίσει πέντε κύριους τομείς πολιτικής. Εγώ σας παρακαλώ να διαβάσετε την έκθεσή μας, γιατί εγώ θα τα πω με λίγα λόγια τώρα. Αν πάρετε το πρώτο από τα πέντε θέματα, η Ευρώπη έχει ανάγκη να συναποτελέσει τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας που να έχει σταθερότητα και κοινή ανάπτυξη. Από αυτό εξαρτάται η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, από τη θέση μας στις παγκόσμιες αγορές και από την συμμετοχή μας στη σταθερότητα και στην ευημερία. Αν εξετάσετε τώρα την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του εμπορίου, βλέπετε προσεγγίσεις σε περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες που δεν θεωρούνται από πολλέ φτωχές χώρες του κόσμου ότι είναι προς το συμφέρον τους. Δηλαδή πάνε εμπορικές πολιτικές και αποσχίζονται από τις οικονομικές πολιτικές. Τελικώς καταλήγουν σε βάρος και της Ευρώπης. Προκαλούν αιμορραγία πόρων από την υποσαχάρια Αφρική. Σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε με ευθυγραμμισμένες πολιτικές. Άλλο θέμα. Κλίμα που ανέφερε πριν ο προλαλής σας κύριος Λανταμπούρου. Η Ευρώπη έχει από τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακος. Έχει μάλιστα και αξιόπιστο ιστορικό σε ορισμένες διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Εκεί όπου δεν έχει αξιόπιστο ιστορικό είναι στην εσωτερική της πολιτική. Μπορεί να κραδένει αυτό τον στόχο του 30% μείωσης του διοξιδίου του άνθρακος, ενώ ταυτόχρονα το ε, σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών είναι στα 5 δολάρια τον τόνο, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλά. Πώς θα ζητήσει υποστήριξη από υποσαχάριες χώρες της Αφρικής σε αυτά. Άλλος τομέας, οι συγκρούσεις. Εμείς που κάνουμε έρευνα για την ανάπτυξη γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι σε μια ζώνη φτώχειας κάτω από ένα εισόδημα λοιπόν που σημαίνει φτώχεια ζουν σε ζώνες και χώρες όπου γνωρίζουν συγκρούσεις. Εκεί μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει καλό ιστορικό διαμεσολάβησης για την ειρήνη, όπως για παράδειγμα στις Φιλιππίνες και στο Ανατολικό Τιμόρ. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές όπου η προσέγγιση μας σε ανθρωπιστικά θέματα αποσυνδέεται από την αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις. Και γνωρίζουμε ότι οι χώρες όταν πια ξεφεύγουν από τη σύγκρουση είναι πάρα πολύ ευάλωτες και μπορεί να ξαναπέσουν σε συγκρούσεις. Εκεί χρειάζεται λοιπόν μια ξεκάθαρη ανθρωπιστική ατζέντα και βοήθεια για την ανοικοδόμησή τους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά μέρη του κόσμου όπου η εξωτερική πολιτική κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση από τις πολιτικές ανάπτυξης και από την ανθρωπιστική υποστήριξη και την, από, την ανοικοδόμηση μετά από συγκρούσεις. Σε άλλο κρίσιμο τομέα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, όπου βεβαίως στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μέσα από τις συνθήκες που οδήγησαν στη γέννησή της έχει πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι αξίες που θα πρέπει να προβάλλει με ένταση στην παγκόσμια σκηνή Ορισμένε φορέ τα καταφέρνει καλά. Σε άλλε δεν τα καταφέρνουμε καθόλου καλά. Για παράδειγμα στην Αίγυπτο, όπου στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα παρισέφρισαν στις ανθρωπιστικές, στον ανθρωπιστικό προβληματισμό, στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Υπάρχουν χώρες που τα καταφέρνουν στην ανάπτυξη, παρόλα αυτά δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι οι αξίες αυτές να προβληθούν σε όλο το φάσμα των πολιτικών μας. Από τις αντιπροσωπείες μας στις διάφορες χώρες, το ίδιο με την προσέγγισή μας σε ε, συμφωνίες επενδύσεων και παντού αλλού. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι η φτώχεια και η ανισότητα. Από την αρχή της ομιλίας μου είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ανθούσα και πιο ισοδίκαιη εξέλιξη στο παγκόσμιο, στην παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Αν εξετάσετε τις σημαντικές, τη σημαντική πρόκληση της μείωση της φτώχειας, υπάρχουν πολλοί τομείς όπου τα καταφέρουμε καλά. Μειώνονται όντως οι αριθμοί των φτωχών. Μειώνεται η θνησιμότητα των παιδιών, νηπίων και βρεφών. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι ο ρυθμός της πρόοδου αυτής μειώνεται και ότι πολλοί άνθρωποι μένουν στην άκρη του δρόμου. Πρόκειται για μια παγκόσμια έκφραση ενός προβλήματος που διαπιστώνουμε και στην Ευρώπη. Πολλά από τα σημεία της συνθήκης της Λισαβόνας αλλά και άλλα νομικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουν ώστε η Ευρώπη να είναι ο σημειοφόρος της αντιμετώπισης όχι μοναχά της απόλυτης φτώχειας, αλλά και της ακραίας ανισότητας σε τομείς όπως η παιδεία, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κλπ. Είπα από την αρχή ότι το πρόβλημα που μας απασχολεί στην έκθεσή μας είναι μια πρόκληση διακυβέρνησης. Συμφωνώ με πολλές από τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Λανταμπούρου, αλλά αυτό που επιθυμώ, αν μπορώ να μιλήσω ευθέως, να πω είναι ποιες είναι ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές της διακυβέρνησης, της χρηστής διοίκησης. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα της σύγκλησης, δεν είναι τίποτε το νέο. Υπάρχει μια δομή διακυβέρνησης που στοχεύει στην ουσία σε μια παραγωγή ανισότητας. Και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Ο στόχος της ε, υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων από την ίδρυσή της ήταν να διαμορφώσει μια ομοιόμορφη εξωτερική πολιτική. Και όμως έχουμε αποκλήσεις ανάμεσα στην Προεδρία και στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Έχουμε 28 Ευρωπαίους Επιτρόπους, οι οποίοι συντονίζονται με αδύναμο τρόπο, δεν προχωρούν στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης ατζέντα της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Άλλη πρόκληση λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά. Η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχευσε ιδίω στην διεύρυνση και στην ασφάλεια. Το δικό μας επιχείρημα που προβάλλουμε στην έκθεσή μας είναι ότι χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό συντονισμό κάτω από ένα πυρήνα επιτρόπων του εμπορίου, των ανθρωπιστικών, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Διότι η αποτελεσματικότητα της Ευρώπης έχει μειωθεί στην παγκόσμια σκηνή. Μιλούμε για μια μετακίνηση στην πολιτική νοοτροπία και αν καταφέρουμε να επιτύχουμε τη μετακίνηση αυτή νομίζω ότι τότε θα ενισχυθεί μάλιστα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συγκρατήσει ενωμένη αυτή την ομάδα πυρήνα των επιτρόπων. Θα τα δείτε όλα αυτά στην έκθεσή μας και θέλω τελικά να απευθύνω μια έκκληση προς εσάς όλη την Επιτροπή Εξωτερικών, διότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καταραίει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1 τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο τρίτα δεν έχουν εμπιστοσύνη. Χάνουν την εμπιστοσύνη του όταν βλέπουν του θεσμού να μην αποδίδουν. Χρειάζεται λοιπόν να αρχίσουν να αποδίδουν στην παγκόσμια σκηνή. Και θεωρούμε ότι εάν οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουμε στην έκθεσή μας υιοθετηθούν, θα αρχίσουν να αποδίδουν και θα επιτευχθεί αυτό που λέμε στον τίτλο μας, δηλαδή να δώσουμε παγκόσμιες λύσεις και να βάλουμε την Ευρώπη στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις εκθέσεις σας. Θα, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή αρχών και στο μέλλον. Και στην έκθεση αυτή θα βρούμε υλικό που θα χρειαστούμε για την ακρόαση. Με την μελλοντική υπατή εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο, για να αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε διάμακρον. Έχουμε χρόνο το πολύ μέχρι 7 παρατέταρτο. Και μάλιστα έχω τώρα 6-7 ομιλητές. Ένα λεπτό ο καθένας. Ή να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία του προπολογισμού. Όχι, είναι στις 12. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με ένα λεπτό. Η κυρία Πλίνσκι. Α, βρίσκεται εκεί. Α, ο κύριος, ο κύριος Πλίνσκι. Είμαι... Νέος... Βουλγαρία. Νέος ευρωβουλευτής από το Euronest. Σε μισό λεπτό μόνο, πρόεδρε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Ανταμπούρ. Το σημείο παραθυμών 5 που μας εξήγησατε σε σχέση με την πολιτική γειτονία σας. Γι' αυτό σας ρωτώ. Με την εταιρική σχέση προς Ανατολάς τι γίνεται. Λέγατε ότι η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε αποδεκτή, δεν ήταν επιστική, γιατί δεν ήταν επαρκής. Για να δώσει κάποιες προοπτικές ρεαλιστικές σε αυτές τις χώρες ούτως ώστε να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε αυτή την εταιρική σχέση που Ανατολάς. και να υπάρξει κάποια συνεργασία με τις χώρες που είναι ακόμα πιο ανατολικά από τις χώρες που ονομάζουμε χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης αντί να προσπαθούμε να τις προσελκύσουμε και έτσι τις χώρες αυτές να τις ε, απομακρύνουμε από τους ε, ακόμη προς Ανατολάς γειτονές τους. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι. Χαίρομαι που με τον κύριο Λανταμπούρου, τον ξέρουμε για 20 χρόνια. Ναι, ναι, είμαι θαυμαστή σα κύριε Λανταμπούρου. Και ο Κέβιν είναι εδώ και οι δύο νομίζω έχετε θέσει πολύ αισιόδοξου στόχου, φιλόδοξου στόχου, αλλά είστε και λίγο αρνητικοί. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποτύχει. Ε, Πέτυχαμε κάποια πράγματα, αποτύχαμε σε άλλα, δεν είναι το πιο δίκαιο. το πρόβλημα τη διακυβέρνηση είναι στην καρδιά των ε, προκλήσεων. Αλλά από την άλλη μεριά, αν λύσουμε δύο προβλήματα, θα δημιουργηθούν άλλα, ίσως περισσότερα. Και όσον αφορά αυτό το μεγάλο κατάλογο των προσφορών, θα μπορούμε να δώσουμε πολιτικό ρόλο στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με τα περισσότερα που μα είπατε. Α πούμε, όσον αφορά τι δυνατότητε άμυνα ή τη διεύρυνση, τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο, αν υπάρχει πολιτική βούληση, νομίζω. Επίση, ε, της, το πολυμερές πλαίσιο διαπραγματεύσεων, ε, ας πούμε στα εμπορικά, ε, δεν μας το είπατε γιατί νομίζω ότι εκεί μπορούμε πολλά να πετύχουμε. Είπατε ότι ε, πολλά θέματα σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και με τη δική μας πολιτική, αυτό είναι καλό. Αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε να υπάρχει κάτι σαν ελάχιστος κοινός παρονομαστής, εξίσωση προς τα κάτω κατά κάποιο τρόπο. Πάντως εγώ διάβασα όσα μας διαβιβάσατε με καλή προσοχή και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας μιλήσετε. Η επόμενη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Νίτς και εγώ, να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Λανταμπούρου. Πρώτα 15 ετίες είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας γιατί τότε προετοιμάσαμε την διεύρυνση. Και είχαμε πάει πολλές φορές στις τότε υποψηφίες χώρες και σήμερα κράτη-μέλη. Μάθαμε πολλά. Πρόκειται για ένα μάθημα πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το να προσπαθεί κανείς να μην απαιτεί από τους άλλους κάτι το οποίο ο ίδιος δεν καταφέρνει να επιτελέσει. Κάτι σαν ε, σεμνότητα, αναγνώριση των ορίων, των ε, μείων εκτιμάτων. Αυτό είναι πιο ενθαρρυντικό παρά να αερολογεί κανείς και να... Είναι πράγματα δυσνόητα. Επομένως, εάν θέλουμε να πετύχει η πολιτική μας σε σχέση με τις τρίτες χώρες, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προβάλλουμε το θέμα της νομιμότητας. Δηλαδή, να είμαστε πιο δίκαιοι, να μην θεωρούμε ότι εμείς από καθέδραση είμαστε τέλειοι και τους τα μαθαίνουμε όλα. Και εμείς δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα. Τελευταία παρατήρηση, για να είμαι σύντομη, ότι οδυνηρά μάθαμε το καλοκαίρι το πόσο τα θεσμικά όργανα είναι αποδοτικά όταν όλα πάνε καλά. Και επίσης ότι τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα, ε, τότε δεν πάρει πάρα πολύ καλά τα θεσμικά όργανα. Ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο ισχύει και όταν έχουμε κάποια κρίση. Τότε φαίνεται πόσο δύσκολο είναι κανείς κάτι να κάνει και πώς μπορεί να βρεθούν κάποιες λύσεις ε, αποτελεσματικές στα δύσκολα. είναι πολύ αδύνατο αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα συγκεκριμένα προβλήματα δεν βρούμε απαντήσει. Muchísimas gracias. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζιγκλέσιας. Πάρα πολύ χαίρομαι που σας αρέσει ο τραγουδιστής και οι τραγουδιστές που ονομάζονται Εγκλέσιας όπως και εγώ. Όντως, αξίζει κανείς να προβληματιστεί, να σκεφτεί και τι έχουμε ακούσει από τους σοφούς ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή, ο κόσμος αλλάζει. Δεν επηρεάζει το γίγνεσθε η Ευρώπη χρειαζόμαστε. επομένω μια ευρωπαϊκή πολιτική που να μπορεί να είναι επιδραστική. Μην είμαστε γίγαντες οικονομικό, να είμαστε στρατιωτικό, πολιτικός. Οπότε τώρα έχουμε καινούργια προβλήματα όπως ο φονταμεταλισμός, οι Ρώσοι που ξανά γίνανε Ρώσοι, πείνα, ε, προβλήματα με το περιβάλλον, προβλήματα αναδυναμιστού πλούτου. Τι φταίει. Φταίει το ότι δεν υπάρχουν οι ηγέτες, δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει συνέπεια σε σχέση με την ε, διακυβέρνηση. Μα τι λέτε. Μπάς και το πρόβλημα είναι ότι λείπει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Μα είπατε για το Μάστριχτ. Αλλά τι έκανε το Μάστριχτ. Έφτιαξε α πούμε την κεντρική τράπεζα ε, χάσανε, χάσαν δηλαδή η κυριαρχία εθνική τα κρατη Και βασικό εργαλείο, όπως είπατε για εργαλεία, είναι να έχουμε μία τρόικα που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θέλουν οι λαοί. Λοιπόν, η δημοκρατία είναι άσχετο με τα προβλήματα που έχουμε εδώ και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ κρατήστε το ένα λεπτό, απαντώ όμως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αποδίδει λόγο ανατρίμηνο στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Φωτίγκα. Κύριε Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή σας. Εγώ το συνοπτικό σημείωμα πρόλαβα να διαβάσω μόνο. Πάντως θεωρώ πως κάποια πράγματα δύσκολα μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς παρά το δίδαγμά σας. Παραδείγματος χάρη, η ανάγκη αναθεώρησης ε, της ε, πολιτικής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής του 2003. Αυτό το χρειαζόμαστε. Η παρατήρηση σχέση με την σύνδεση ή και τη διεύρυνση είπατε ότι ε, δεν είναι τόσο σεξι όσο στη δεκαετία του 90 δεν είναι τόσο ελκυστική. Ε, πάντως αυτά που είπατε μόνο μία φορά άκουσα να μιλάτε για αλληλεγγύη. Όταν ε, μιλήσατε για την ανάγκη αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης Και επίσης ε, αναφερθήκατε στις περιοχές ε, όπου από γεωπολιτικής πλευράς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και απαιτείται μια κοινή προσέγγιση από πλευράς μας. Η νεοεμπειραλιστική πολιτική της Ρωσίας ε, δεν είναι στον κατάλογο που μας παρουσιάσατε. Όταν βλέπουμε την πολιτική της Ρωσίας, κυρίως σε σχέση με την Ουκρανία, δεν συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται για ένα μόνο παράδειγμα μιας πολύ συγκεκριμένης ειδική συνεκτικής και σφαιρικής ρωσικής πολιτικής σε σχέση με όλες τις ε, γειτονικές χώρες, τις χώρες με τις οποίες ε, συνορεύει και σε ένα ορισμένο βαθμό με κάποιες χώρες της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ή χώρες του Νότιου Κάφκασου. Για κάποιες χώρες δεν είναι τόσο ελκυστική πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι τις έχει εγκαταλείψει η ευρωπαικη ενωση θεωρουν οτι θα Ένωση. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ συγκεκριμένοι. Ίσως ε, η βαθύτερη ενοποίηση δεν είναι η λύση για να αντιμετωπίσουμε τις εστίες έντασης σε αυτές τις περιοχές. Η κυρία Γκόμες, ε, κύριε Λανταμπούρο, κύριε Βότκινς, ε, συμφωνώ πάρα πολύ με όλα αυτά που είπατε. Η ανισότητα είναι κεντρικό ζήτημα. Δεν πρόκειται μόνο για το πώς διευρύνεται αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για το εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Είναι θέμα δημοκρατίας. Το θέμα της φοροδιαφυγής ε, είναι άλλο κεντρικό ζήτημα. Κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό, αλλά δεν αναφερθήκατε σε αυτό, είναι τα πυρηνικά όπλα και η πυρηνική ενέργεια. Πώς θα είμαστε αυτάρκεις ε, ενεργειακά αν δεν ασχοληθούμε και με την πυρηνική ενέργεια. Πέρα δηλαδή από το, ε, την πτυχή της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας υπάρχει το θέμα της ενεργειακής αυτάρκειας. Τώρα για τη συνοχή της εξωτερικής μας πολιτικής. για την κοινή πολιτική άμυνας και κοινή εξωτερική πολιτική έγινε μια απόπειρα να είμαστε ε, συνεκτικοί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά μπορεί να πει κανεί, τέλο πάντων έγινε προσπάθεια. Όμω, εάν δεν συνεκτιμήσουμε και τα θέματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, και συγκεκριμένα την ε, τροποποίηση, τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της δικής μας εκπροσώπησης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι είναι δυνατόν να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Είμαι ένα πραγματικό μέλος της Επιτροπής ε, και Αντιπρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης. Είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση. Την καλωσορίζουμε και όντως ο Παγκόσμιος Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί όπου έχουμε ήδη ηγετικό ρόλο. Εμπόριο, ανάπτυξη και περιβάλλον. Και όντως χρειάζεται συντονισμός, διότι να αλληλένδεται αυτή η τομή. Ο κύριος σε μίλησε για την ανάγκη συντονισμού και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι ήδη σε αυτή την Επιτροπή για αρχή θα μπορούσαμε να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε συνεργασία με ε, συναρμόδιες επιτροπές. 50 δευτερόλεπτα μίλησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα συντομότατο ερώτημα προς τους δύο προσκεκλημένους μας. Ε, παραπέμπω σε μία δήλωση του κ. Γιούνκερ που μας είπε ότι την επόμενη πενταετία θα ε, πάυσει οποιαδήποτε διεύρυνση, διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική επίπτωση αυτών των δηλώσεων ε, στις βαλκανικές χώρες ή σε όποιες χώρες εργάστηκαν ε, σκληρά για να ε, φέρουν σε πέρας μεταρρυθμίσεις όπως η Μολδαβία ε, θα είναι ανυπολόγιστες. Έπονται και σε αυτή τη χώρα. Για την Μολδαβία λοιπόν ποια θα είναι οι επιπτώσεις των δηλώσεων του κυρίου Γιούνκερ για τον πληθυσμό αυτής της χώρας. Ένα λεπτό μου είπατε και ήσασταν και πολύ σοβαρός, θα το σεβαστώ. Συμφωνώ με αυτά που υπονοείτε στις ερωτήσεις σας. Όντως ε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ε, να ε, δρούμε αλληλέγγυα, να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, αλλά να έχουμε ένα φιλόδοξο ρεαλισμό ως άξονα γνώμονα. Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου δεν χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν λόγω της αποτυχίας των κυβερνήσεων. Έχουμε γίνει πολλές συζητήσεις για την Ουκρανία και τη Ρωσία και δικαίω, αλλά ε, και το Μάλι, το Νότιο Σουδάνι, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εκεί η αποτυχία σφαιρικής προσέγγισης, αφενός δηλαδή ε, θεματολόγιο εξωτερικής πολιτικής, ανθρωπιστική βοήθεια και αφεντέρου αναπτυξιακή πολιτική, οφείλονται σε αποτυχία των κυβερνήσεων. Ε, ε, χρειαζόμαστε ο όντως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα δίκτυο ε, ενοποιημένο για τον άνθρακα παραδείγματο χάρη ε, θα ήμασταν πολύ πιο αξιόπιστοι αν είχαμε ένα ενοποιημένο δίκτυο και συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης Χρειαζόμαστε μια έκθεση όπου θα αναφέρουμε όλες αυτές τις φιλοδοξίες και να στάξουμε ε, από κοινού όλες τις συναρμόδιες επιτροπές αυτές, ε, αυτό τον κατάλογο ε, φιλοδοξιών που έχουμε, των στόχων. Ε, οι στόχοι και οι πολιτικές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν υιοθετήσουμε και μια διαφορετική προσέγγιση για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση. Και σωστά τα είπε ο κύριος Χάουιτ, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε σαν να ήταν ιδανική η κατάσταση. Όχι, ας είμαστε ρεαλιστές και στην εμπορική πολιτική ε, για την ατζέντα μετά το 2015 να δούμε σε ποιους τομείς μπορεί να καθιερωθεί ως ε, ε, ε, να ο, εταιρικό, ο, συγγνώμη, ο ηγετικός ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορίστε και δεν ξεπέρασα και πολύ το χρόνο μου. Και εγώ, λέει ο κ. Λαταμπόρ, θα απαντήσω σε ένα λεπτό. Βλέπω ότι σημαντικές διαστάσεις απόψεων δεν υπάρχουν σε σχέση με τα πορίσματα του μανιφέστου μας. Ε, είπε ο κύριος Χάουιτε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ε, η πολιτική βούληση να ακολουθήσει σωστή κατεύθυνση. Πώς να εκφραστεί αυτή η πολιτική βούληση. Ξέρετε, ε, τα θεσμικά όργανα, είτε μιλάμε για την Επιτροπή είτε για το Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να προβαίνουν σε ε, ε και ε, ε, αναλύσεις της, κατάστασης, της κατάστασης, ούτως ώστε, όπως είπατε κύριε κύριε να ε, γνωρίζει ο λαός τι γίνεται, αλλά το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και για, την, ε, ε, για τις κυβερνήσεις, ώστε να υπάρχει και η όθεση για τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ή να υπάρχει ο προβληματισμός για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεύτερον, εκεί πέρα που θα έπρεπε να έχουμε ισχυρότερη βούληση για την ισχυρότερη ενοποίηση, είναι ακριβώς οι συζητήσεις και οι προτάσεις που γίνονται όχι μόνο από τους επαϊόντες των Think Tank, όχι, και στα θεσμικά όργανα και στις χώρες σας και στα κόμματα. Μιλάτε πολύ στα, στα κόμματα, μιλάμε, μάλλον να το πω στον πρώτο πολιτιστικό, γιατί και εγώ είμαι μέλος κόμματος, ε, μιλάμε στα κόμματά μας για την Ευρώπη αρκετά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, που θα... Ε, λειτουργήσουν ως εφαλτήρια για τις νέες πρωτοβουλίες. Έτσι προχωρούσε ανέκαθεν η Ευρώπη επί τη βάση ιδεών γυναικών και αντρών που έκναν ότι να έχει έρθει η σωστή χρονική στιγμή για να προχωρήσουμε. 1,56 στα Ισπανικά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω για το ότι η Τρόικα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία πολιτικής. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Ε, το κοινοβούλιο είναι το σημαντικό. Γιατί έτσι κάνουμε μια καρικατούρα. Αμαυρώνουμε την εικόνα της Ευρώπης και βλέπουμε ότι όλα είναι αρνητικά. Όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Θέλουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι να είναι ισχυρή η Ευρώπη για να ε, υπεραμεινθεί των ε, αξιών που πιστεύουμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή και την δημοκρατία. Πρόεδρος. Ο πρόεδρος Μπροκ. Ευχαριστώ ε, τους δύο κυρίους. Όπως είπα και πριν, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση με το ευρύ περιεχόμενο. Να δούμε και πώς μπορεί ίσως να μεταφραστεί εντό εισαγωγικών σε ένα κατάλογο πολιτικών ετοιμάτων. Να εξεύρουμε μέσα από αυτήν το υλικό για να φτιάξουμε και μια έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών. Η εξωτερική πολιτική ούτως ή άλλως εξαρτάται σε μέγα βαθμό από τις ε, άλλες πολιτικές και του κλίματος και εμπορικές και αναπτύξεως. Ίσως λοιπόν αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο των εκθέσεών σας είναι πολύ σημαντικό και για την περαιτέρω δική μας εργασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Θα παραμείνουμε βεβαίως σε επαφή. Thank you for IMEC, yes. Uh, we will appreciate Now let's read it. Ciao. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έρθουμε τώρα στο θέμα του προϋπολογισμού. Θέλουμε να ψηφίσουμε αύριο στις 12. Από πλευρά του εισηγητού υπάρχουν παρατηρήσεις. Herr Balz. Κύριε Παλσίτης, εκεί είστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα πεντάλεπτο μας μένει από ό,τι γνωρίζω. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα σπουδαίο, απλώς να ευχαριστήσω όλους. Όλους, συντονιστές, σκιώδεις συγητές, εκπροσώπους πολιτικών ομάδων και έχω κατεβάσει 56 τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να περικόψω τις περικοπές του Συμβουλίου. Συζητήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζυγίσουμε μία μεριά το τι θέλουμε να πετύχουμε και από την άλλη τι ε, χρηματικούς πόρους έχουμε διαθέσή μας. Ε, είναι οι προθέσεις μου αυτές, ε, αλλά έχω συγκεράσει από τις δικές μου με τον άλλον σαν από τα άλλα κόμματα. Και έτσι πιστεύω ότι ήταν σωστό το ότι συμβαστήκαμε για κάποια δύσκολα ζητήματα. Ας πούμε, ο κύριος Πρέντα έχει υποβάλει σχετικά την ε, ε, τροπολογία 11 για την ε, αντιπροσωπεία στο Ιράν. Επίσης πιστεύω ότι θα τα βρούμε σε κάποια επόμενη συνεδρίαση. Η συνάντησή μας δεν συμφωνώ με την τροπολογία Λέζινγκ για να σταματήσει η χρηματοδότηση της αστυνομικής αποστολής στο Κωσυφοπαίδιο και να κλείσουμε ε, την ε, υπηρεσία της Frontex και να στείλουμε ε, πολιτικούς υπαλλήλους. Όχι, εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται πόροι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Επίση, έχουμε δύο τροπολογίες της χώρες της Μεσογείου, ο κύριος Πρέντα συμφώνησε και ο κύριος Μίτσοκ όσον αφορά παραπάνω διάθεση 10 εκατομμυρίων για την Παλαιστίνη. Ε, σύμφωνα με την πρόταση Σάκη, όσον αφορά το 5-0-1-1-1 και 1 και 2 για την Δυτική Σαχάρα, την Παλαιστίνη, ε, γιατί χρειάζεται σε αυτά τα κονδύλια να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Οπότε, παρακαλώ αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν τις τροπολογίες να μου πούν ποιοι θα αναλάβουν να κάνουν τι. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτέ τι τροπολογίε. Επίσης, για αυτό το κέντρο μελετών στην ε, Ουκρανία, στο Χάρκοβο, υπευλήθη κάποια πρόταση να αλλάξει η ονομασία ότι θα πρέπει να ονομάζεται κέντρο μελετών για Ρωσία και Ουκρανία. Εάν συμφωνεί η κυρία Χάρμς για αυτές τις μικρές αλλαγές, σε αυτή την περίπτωση, εντάξει. 5094. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl... Συνεχίζω κύριος Αυτά κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να πω κάτι άλλο σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού για το 2015. Πρίδα. Το λόγο στον κύριο Πρέντα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αμέσω μετά πρόκειται να συνεδριάσουμε οι σκιώδη ηγητέ για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό, ιδίω για το θέμα των πόρων για το Ιράν ε, ε, δύσκολο σημείο. Επίσης, εμείς ξεκινήσαμε από το ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής πρικοδότηση και χρηματοδότηση. Να εξασφαλίσουμε ότι οι πιο σημαντικές προτεραιότητες θα καλυφθούν. Και η αντιμετώπιση, ξέρετε, των κρίσεων είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί οι κρίσει δεν θα λιγοστέψουν, θα αυξηθούν, άρα δεν πρέπει να υπάρχουν λιγότερα χρήματα για αυτέ τι κρίσει από ό,τι πριν. Επομένω, είναι το θέμα επίση των παρατηρητών των εκλογών. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη, τα κονδύλια του 2014. Κατά τριτών δε, έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα. Μας ενδιαφέρουν, είναι προτεραιότητες. Και έχουμε και την πρόταση Γκάλερ για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Άλλο πρόγραμμα το οποίο το είχε προωθήσει ο κύριος ε, Φράγκα όσον αφορά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Νότιο Κεντρική Αμερική και εσεί κύριε Πρόεδρε έχετε ένα δικό σας πρόγραμμα για την ε, διαδικασία του μετασχηματισμού και τη μεταβατική περίοδο του πάντων στις σχέσεις μας με την Λευκορωσία. Όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλιστούν, να καλυφθούν. Ελπίζω ότι θα τα βρούμε και αύριο στην ψηφοφορία δεν θα διχαστούμε. Και βλέπετε πώς θα που κοιτάω, προς τον συνάδελφο Howitt. Γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια θεματάκια που δεν έχουν επιληθεί με εκείνον. Νομίζω ότι, λέει κύριε είναι τώρα η ώρα να δούμε τις προτεραιότητες. Γιατί είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα το πού θα πάνε τα χρήματά μας. Έχουμε στη γειτονιά μας γύρω-γύρω κρίσεις. Ένα σωρό. Μην το ξεχνάμε. Επίσης, είναι προτεραιότητα η πολιτική γειτονία προ Ανατολά. Και είπαμε επίση να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην Παλαιστίνη, μια που η κατάσταση τόσο έχει δυσκολέψει εκεί. Χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και επίση να σα ευχαριστήσω όλου συνάδελφοι για τη συνεργασία μαζί σα. I was going to remain silent, but I can't uh, help but make a short intervention after our friend. Ήθελα να σιωπήσω, αλλά μετά από αυτό που ο κύριο Πρέντα δεν μπορώ. Και θα μιλήσω έστω και σύντομα. Πρώτα πρώτα φορά τον κύριο Μπαλτσίδη, το πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, ήταν μεγάλη, δύσκολη η πρόκληση αμέσω μετά τι εκλογέ. Γρήγορα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αλλά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και είμαι σίγουρο ότι θα βρεθούμε και θα τα βρούμε. Συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται για τα χρήματα για την προσωπία στο Ιράν, εμείς θέλουμε να υπάρχει εκεί μια μόνιμη αντιπροσωπεία στη χώρα. Και σέβομαι τη στάση, τη θέση του ΕΛΚ. Και θέλουν δηλαδή να περιμένουν να δουν πού θα πάνε οι ομιλίες με τη χώρα, με το Ιράν. Τώρα βέβαια ο καθένας δίνει άλλο περιεχόμενο στην έννοια επιτυχία. Εμείς πάντως αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις με το Ιράν και έτσι να έχουν ο τέλος οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Να, κάναμε τη χειρονομία αυτή για το ΕΛΚ. Να μην ψηφίσουν κατά, να, να απόσχουν. Και έτσι να τα βρούμε. Και εμεί να κάνουμε το ίδιο με τι δικέ του ε, τροπολογίε και έτσι να περάσουν οι τροπολογίε. Όμω να μην καταψηφίσει το ΕΛΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραία πρόταση συμβιβαστική. Θα χαρώ πάρα πολύ αν κλείσει μια τέτοια συμφωνία συμβασμού. Well, uh, unsurprisingly, um, the ECR group is opposed to any δεν θα σας εκπλήξω. Εμείς είμαστε κατά οποιασδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού για, σε, για την εξωτερική δράση. Πιστεύουμε ότι μπορεί να περικοπεί έτσι περαιτέρω ε, προϋπολογισμό στα πλαίσια της λιτότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Γενική Αρχή. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε έκκληση για αύξηση του προϋπολογισμού και ξαναλέω πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν και περικοπές. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν και κάποιοι έκτακτοι τομείς, όπως είπαν και οι συνάδελφοι για την ανατολική γειτονία, η ε, ανατολική εταιρική σχέση, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με αυτά που τώρα συμβαίνουν στην Ουκρανία, ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο, Αφρική και Ιράκ, ε, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσαρμογές στο προϋπολογισμό εν γέννη, όμως θα υποστηρίξουμε την πρόταση του Συμβουλίου για περικοπή. Ε, για το θέμα του Ιράν είναι πολύ λεπτό το ζήτημα ε, και είναι ισχυρή επιχειρηματολογία και των δύο πλευρών. το, η πολιτική μου ομάδα πιστεύει ότι δεν έχει οριμάσει ακόμη ο, ε, η στιγμή δεν ε, είναι σκόπιμο να είναι την προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Ε, φυσικά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και μπορεί σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν τώρα στο Βόρειο Ιράκ για την καταπολέμηση των μαχητών του Ισλαμικού κράτους να χρειαστεί να αλλάξει η κατάσταση. Πάντως αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να συντρέχουν προϋποθέσεις όπου θα πρέπει πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας. Ε, πάντως προς το παρόν ε, δεν ε, παρκούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις του Ιράν ώστε να πιστούμε για το ότι έχουν εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό τους πρόγραμμα ώστε εμείς να δεχτούμε οτιδήποτε που η Τεχεράνη θα εκλάβει ως βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Το θέμα των προτεραιοτήτων αναφέρθηκε από διάφορους συνάδελφους. Κατά τη γνώμη μας, ο προϋπολογισμός γίνεται λένε και πιο αδιαφανής και η ε, προτεραιότητα κατευθύνονται προς περαιτέρω στρατιωτικοποίηση, περισσότερη έρευνα για στρατιωτικό εξοπλισμό και προώθηση ε, ο πολιτικών ε, συμφερόντων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι αυτό επιβαρύνει την αναπτυξιακή πολιτική και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, είναι δυνατόν να γίνουν περικοπές σε τέτοιους τομείς και σε άλλους τομείς να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τις σχετικές τροπολογίες. Θα πρέπει να ε, προβούμε λοιπόν σε περικοπές για τα μέσα που ενδέχεται να ε, οξύνουν ε, τις ε, διαμάχες και, να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους. Φυσικά θα υποστηρίξουμε με οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Πρόεδρος, έμαθα μόλις ότι ε, τα θεσμικά όργανα έχουν, σε ενός αποσταθεροποιητικό ρόλο ε, σε σχέση με τη, τα αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία. Κύριε Πρέντα, θέλετε τι, να κάνετε σχόλιο ε, για αυτό που μόλις είπα. Όχι. Σα. γίνει αύριο η ψηφοφορία. Μόνο υπάρχει μια τροπολογία για το Σαρκίφτο ερευνητικό κέντρο. Για το κέντρο ερευνών. <laughs> Ich äh, bedanke mich sehr herzlich. Wir sehen uns morgen früh 9. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο πρωί-πρωί με την ε, Ιταλίδα Υπουργό Εξωτερικών. 8 η ώρα του διευρυμένου Προεδρείου. Ich schlage diesen Titel vor, Center for Ukrainian and Russian Relations. Yeah. Ναι.